Dear colleagues, shall we start our afternoon meeting? Okay, and then I will continue in Lithuania. Συνεχίσω λοιπόν λιθουανιστή. Ε, ε, Ξεκινάμε λοιπόν την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση και το πρόγραμμά μας που είναι στην ημερήσια διάταξή μας το σημείο 11. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία για τη μητρική άδεια. Θα ανταλλάξουμε απόψεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Η κυρία Βιβίσου εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι εδώ. Έχουμε εκπροσώπους της Λετωνικής Προεδρίας εδώ. Δεν βλέπω να υπάρχουν. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα, γιατί χτες η Λετωνική ε, Προεδρία μας είπε ότι θα στείλει εκπρόσωπο στη συνεδρίασή μας και ότι θα εκφραστεί η άποψη της Προεδρίας. Μόλις μάθαμε ότι η Λετωνική Προεδρία δεν εκπροσωπείται και μάλιστα δεν εκπροσωπείται χωρίς δικαιολογία, είναι αδικαιολόγητα πούσα, κακό προηγούμενο είναι αυτό. Όλα τα θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες της Προεδρίας πρέπει να συνεργάζονται για να πετύχουμε και να πετυχαίνουμε καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Eurofon, τον κύριο George Καπρίτα, που θα παρουσιάσει την αρχική μελέτη για την μητρική άδεια στα διάφορα κράτη-μέλη. Κύριε Ζωζ Καμπρίτα, έχετε το λόγο. Chair, thank you Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ήλπιζα, ήλπιζα να είχα κάποια εικόνα στην οθόνη έχω μια παρουσίαση και κάποιες διαφάνειες να σας δείξω. Ελπίζω οι τεχνικοί αν μ' να ανάψουν τον προβολέα, το μηχάνημα προβολής. Θα ήθελα συνεχίζοντας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και διαβίωσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γυναικών που μας προσεκάλεσε εδώ Βασικός στόχος της παρουσίασής μου είναι να σας παρουσιάσω κάποια αρχικά αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε όσον αφορά τη διατάξεις περιμητρικής αδείας των κρατών μελών της Ένωσης κάτι που ζητήθηκε την Επιτροπή Γυναικών ούτω ώστε να έχετε μια επίκαιρη άποψη σχετικά με αυτό. Κάποια στοιχεία για το όλο ιστορικό για να τα έχουμε υπόψη. Η οδηγία 92 92-85 εξετάζεται σήμερα εδώ εν ώψη ενδεχόμενη αναθεωρήσεω μέτρα για βελτιώσεως βελτιώσεω για την ασφάλεια και την υγεία στον τόπο εργασία των οικείων γυναικών και ε, γυναικών που έχουν γεννήσει πρόσφατα και φυλάζουν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την οδηγία 2010-18 τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που καθορίζει την ελάχιστη διάρκεια της γονικής αδείας στο τετράμινο. Η οδηγία όμως δεν προβλέπει ελάχιστο ποσοστό αντικατάστασης των εσόδων των γονέων που παίρνουν αυτή την άδεια και υπάρχουν άλλα δύο μέσα σημαντικά. Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την Ευρώπη του 2020 υπογραμμίζουν τη σημασία της εφαρμογής εξολογήσεως των πολιτικών περιαπασχολήσεως που προωθούν την ισότητα των φύλων και την ισορροπία ε, ζωής στον τόπο εργασίας και οικογενικής ζωής. 75% επίπεδα προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους στόχους στρατηγικής του 2020. Και έχουμε την οδηγία 2006-54 που είναι η, οδηγία αναδιατύπωσης, recast, και τονίζει ότι τα κάτι μέλη θα ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους να προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών, θα προωθούν ευέλικτες διευθετήσεις για την εργασία για να διευκολύνουν τη συμφιλίωση εργασίας και ιδιωτική ζωής. Για να συνεχίσω πρέπει να κάνω μια διάκριση ε, μεταξύ τριών σημαντικών ορισμών. Όταν μιλάμε για οικογενειακή άδεια, αγωνική άδεια, μετρική άδεια και πατρική άδεια. Μητρική άδεια συνήθως χορηγείται στις μητέρες και σημαίνει ε, ένα διάλειμμα από την εργασία πριν τη γέννα και μετά τη γέννα. Και είναι βασικές περίοδοι για φυσική ανάκαμψη της μητέρας μετά την ιτότα. Η γονική άδεια θεωρείται ότι είναι δικαίωμα των εργαζομένων και στα δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται και είναι διαθέσιμες άδειες και στους δύο γονείς Βασικός στόχος είναι να προσέχουν το νεογέννητο, το παιδί μέχρι κάποια ηλικία. Συνήθως αυτή η άδεια λαμβάνεται μετά τη μητρική, την περίοδο της μητρικής ή πατρικής άδειας. Και έχουμε την πατρική άδεια, την άδεια πατρότητας που δεν καλύπτεται από κάποια οδηγία, δεν υπάρχει ε, νομοθεσία ευρωπαϊκή. Είναι μια σύντομη περίοδος ε, αδείας που χορηγείται στον πατέρα ούτως ώστε ο πατέρας να έχει κάποιο χρόνο να μπορεί να το περάσει με το παιδί και με τη σύντροφό του. Βλέπουμε τρεις διακριτές περιπτώσεις ε, αδείας. Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα είναι η διάρκεια της άδεια μητρότητας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε την πιο, τις πιο σύγχρονες ε, πληροφορίες για τη διάρκεια της αδίας μητρότητας. Είναι ατυχέστατο το ότι δεν έχουμε τη διαφάνεια, διότι θα βλέπατε τότε την απίστευτη διαφορά που υπάρχει μεταξύ κρατών μελών. Και... Α, βλέπουμε την εικόνα. Θα δείτε λοιπόν στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει μια χρονική περίοδος υποχρεωτική και συνολική χρονική περίοδος που συλλαμβάνει την υποχρεωτική περίοδο και ε, ε, εθελοντικές περιόδους που μπορεί να ζητήσουν οι μητέρες πριν γεννήσουν και μετά τη γέννα. Δεν βλέπουμε ακόμα τη διαφάνεια που θα ήθελα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η ακραία περίπτωση που έχουμε στη Σλοβακία, 34 εβδομάδες μητρικής ε, άδειας μητρότητας, υποχρεωτικές ε, εβδομάδες πρέπει να πάρουν οι μητέρες την άδεια για 34 εβδομάδες. Βλέπετε αριστερά. Οι γαλάζιες γραμμές είναι η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας. Οι κοκκινοπές γραμμές δείχνουν το υποχρεωτικό τμήμα της άδειας. Στο άλλο άκρο, στα δεξιά, βλέπετε χώρες όπως είναι η Λιθουανία και η Λετωνία, όπου δεν υπάρχει ακόμα υποχρεωτική ε, άδεια που προβλέπεται από την νομοθεσία τους. Βλέπετε πόσες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ε, διάρκεια. Άλλο σημαντικό θέμα, σε ποιο βαθμό ο μισθός, οι αμοιβέ των εργαζομένων καλύπτονται κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περίοδου. Οι μητέρες παίρνουν την άδεια, πόσο επηρεάζεται το εισόδημά τους, πόσο, πόση απώλεια εισοδήματος καλύπτεται από το επίδομα μητρότητας. Στα περισσότερα κατημέλη, αυτά που είναι πράσινα εδώ, Υπάρχει 100% αντικατάσταση του εισοδήματο. Υπάρχουν άλλε περιπτώσει όπω η Ιρλανδία, γαλάζιο χρώμα. Ε, εκεί έχετε καταποκοπήν ποσό. Δεν υπάρχει άμεσο συσχετισμό με το εισόδημα του εργαζομένου. Και έχουμε μετά τις περιπτώσεις τη τσεχική δημοκρατία της Βουλγαρίας, και Σλοβακίας όπου το ποσοστό αντικατάστασης δεν ξεπερνά το 65% στη Σλοβακία και 70% στη Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία. Συγγνώμη, Αυτό δείχνει επίσης ότι η κάλυψη δεν είναι ομοιογενής σε όλα τα κράτη-μέλη και είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν συζητούμε το θέμα. Άλλο ζήτημα που το εξετάσαμε στην έρευνά μας η ευθύνη για την καταβολή, για την πληρωμή, για την άδεια μητρότητας ποικίλει από χώρα σε χώρα. Οι δημόσιες αρχές και η κοινωνική ασφάλιση είναι υπεύθυνοι φορείς για την καταβολή των πληρωμών του επιδόματος μητρότητας. Σε κάποιες χώρες υπάρχει μείγμα θεσμών, φορέων, στην Αυστρία, στην Ελλάδα, ε, δημοσίου τομέα. Στη Γερμανία έχουμε εργοδότη και ασφάλεια υγείας. Ο εργοδότης πληρώνει ένα τμήμα και ασφάλεια υγείας το υπόλοιπο τμήμα. Δανία, Μάλτα, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί οι εργοδότες είναι υπεύθυνε για την καταβολή αυτής της πληρωμής κατά τη χρονική περίοδο όπου οι εργαζόμενοι έχουν την άδεια μητρότητας. Η Μάλτα είναι η μόνη χώρα που οι εργοδότες φέρουν πλήρως την ευθύνη για την κάλυψη. Δεν υπάρχει κάποιο επίδομα, κάποια αποζημίωση για να βοηθήσει εργοδότες Στη Γερμανία, Ρωμανία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπεύθυνοι εργοδότε η διαβολή του ποσού αυτού, αλλά επιστρέφεται το ποσό της δημόσιε αρχέ, στι κρατικέ αρχέ. Στην Μάλτα γίνονται πρόσφατα συζητήσει για την αλλαγή του καθεστώτος, ούτω ώστε οι εργοδότες να μην έχουν το πλήρε βάρος ε, του επιδόματος μητρότητα. Κάτι ενδιαφέρον από αυτά που είδαμε και από αυτά που μας ζητήσατε ήταν που είδαμε τη σχέση μεταξύ του επιδόματος άδεια μητρότητας ε, και του επιδόματος ε, αναρωτικής ανάρρωσης. Ε, διότι στα 19 κράτη-μέλη δεν σχετίζονται τα δύο, δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ άδεια μητρότητας και του σχετικού επιδόματος και της αναρωτικής άδεια και του επιδόματος του αναλόγου. Ε, παρόλα αυτά Υπάρχει άμεση σχέση από ό,τι είδαμε μεταξύ των δύο. Το είδαμε από τα γραφήματα. Ε, βέβαια όλοι σήμερα γνωρίζουμε ότι η μητρότητα δεν είναι ασθένεια, αντιθέτως είναι σημείο υγείας και δεν πρέπει να θεωρηθεί ή να αντιμετωπιστεί ως ασθένεια. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες χώρες όπως είναι η Τσεχική Δημοκρατία, καταβάλλονται και τα δύο επιδόματα στα πλαίσια του συστήματος ασθεν... ασθενείας. Στην Εστονία η μητρότητα θεωρείται σαν μια προσωρινή αδυναμία να εργαστεί κανείς παρόμοιο φαινόμενο όπως ε, κάτι προξαλούν οι ασθένειες. Στη Φιλανδία ε, καλύπτονται σύμφωνα με, το επίδομα, με την ασφάλεια υγείας, Ουγγαρία και τα δύο καλύπτονται τα επιδόματα από το σύστημα ασφαλείας και, ε, και υπολογίζονται παρομοίως και στο Λουξεμβούργο και αυτό μας εκπλήσει, θεωρείται σαν περίοδος αναρωτική. Για να πάρει κανείς ε, την άδεια μητρότητας χρειάζεται πιστοποιητικό από το γιατρό όπως όταν κανείς ασθενεί στη Σουηδία. Τα επιδόματα μητρότητας αντιστοιχούν στα επίπεδα επιδόματος ασθενείας. Υπάρχει ε, συσχετισμός μεταξύ των δύο. Όμως, συγκρίνοντας τα επιδόματα που καταβάλλονται και από την άδεια μητρότητας και από την πληρωμή για την ανάρρωση, ε, για την άδεια μητρότητας τα επιδόματα είναι πιο γενναιόδωρα. Αλλά σε κάποιες περιστάσεις ε, το επίδομα ασθενείας μπορεί να είναι πιο υψηλό από το αντίστοιχο για την άδεια μητρότητας, οπότε χρειάζεται να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες για να καταλήξουμε σε τελικά πορίσματα. Άλλο που μας ζητήθηκε. Σχετικά με τα άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας περί αδείας μητρότητας, όπου εκεί που αναφέρεται ότι οι έγκες ή θυλάζουσες εργαζόμενες δεν υπέχουν υποχρέωση να εκτελούν εργασίες που απειλούν την υγεία τους και την ασφάλειά τους, να εκτεθούν σε φυσικές ουσίες, χημικές ουσίες, βιολογικές ουσίες ή ε, νυχτερινές βάρδιες. Τι συμβαίνει όμως αν πρέπει να μεταφερθούν σε μια θέση απασχόλησης που πληρώνεται ε, λιγότερο. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους να εκτεθούν σε ουσίες ή συνθήκες που είναι επικίνδυνε για την υγεία τους. Υπέχει ε, υποχρέωση εργοδότης να τις μεταθέσει σε μια άλλη θέση. Τι γίνεται όμως αν εκτελούν μια εργασία που αμείβεται χαμηλότερα. Στις περισσότερες χώρες και στα περισσότερα κάτι μέλη εν γέννη, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εισπράττουν ένα ποσό που ισοδυναμεί με το μισθό τους πριν την εγκυμοσύνη αν η προσαρμογή που γίνεται σε νέα θέση είναι κάτι ανέφικτο, στις περισσότερες περιπτώσεις τους χορηγείται ένα επίδομα που αντιστοιχεί ε, στην άδεια μητρότητας. Οπότε υπάρχει μια ανάκτηση του εισοδήματος. Σε κάποιες χώρες πρέπει να πάρουν τη χαμηλότερη αμοιβή, αλλά μετά υπάρχει μια αποζημίωση, ένα επίδομα που καταβάλλεται από τις δημόσιες αρχές και έτσι γεφυρώνεται διαφορά μεταξύ των όσων εισέπραταν πριν και ό,τι έπραταν κατά τη διάρκεια τη προσωρινής περίοδου διότι δεν μπορούσαν να εκτίθενται σε διάφορες περιστάσεις που σας περιέγραψα προηγουμένως. Αυτά που περιγράφουν τα άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας. αλλα κάτι κράτη-μέλη, και αυτό είναι σημαντικό, είναι σαφέστατο ότι από την νομοθεσία. Την εργατική νομοθεσία λέγεται ότι επουδενή εργαζόμενη εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να κερδίζουν λιγότερα από αυτά που κέρδιζαν πριν να είναι έγκυες αυτές οι γυναίκες πριν ξεκινήσει η εγκυμοσύνη τους. Αυτό ισχύει στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Ε, κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω εκτενέστερα, ίσως αργότερα, αφού παρέμουν οι άλλοι συνάδελφοι, είναι και το εξή. Η άδεια μητρότητα πρέπει να ειδωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ένα σύστημα αδειών. Άδεια μητρότητα, άδεια πατρότητα, ε, γονική άδεια, όλα αυτά είναι ένα περίπλοκο σύστημα, ένα σύνολο ε, που σχετίζεται με διάφορες αποφάσεις προσλήψη στις περισσότερες ε, περιπτώσεις στον επίπεδο νοικοκυρίου πρέπει να ληφθεί η απόφαση. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν χώρες με ελάχιστη ή μη πρόθεση του ρόλου του πατέρα. Δεν υπάρχει άδεια πατρότητας. Υπάρχει γονική άδεια, αλλά είναι άνευ αποδοχών και μετά υπάρχουν διάφορες καταστάσεις όσον αφορά την άδεια μητρότητας. Διάρκεια, διαφέρει, η αμοιβή διαφέρει. Το θέμα είναι ότι βασικά το βάρος ε, είναι στους ώμους των γυναικών περισσότερο ή μάλλον αποκλειστικά αλλά δεν είναι οι μόνες υπεύθυνε για τη γέννηση του παιδιού και το παιδί. Έχετε τις μητέρες, τους πατέρες, οπότε υπάρχει ανισορροπία. Αυτό μπορούμε να το δούμε αργότερα. Τι τονίζω, ότι θα πρέπει να θεωρηθεί η άδεια μητρότητα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Όπως κάποιοι λένε μέσα σε ένα περίπλοκο σύμπλεγμα αδειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι τρεις προαναφερθήσεις άδειες. Και άλλες σημαντικές πτυχές θα ήθελα ακροθυγώς να σας αναφέρω. Αυτό που είδαμε είναι ότι οι εθνικές έναμες τάξεις επηρεάζουν τα πράγματα. Αν υπάρχουν υποχρεωτικές άδειες που πρέπει να ληφθούν, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά ε, το να ζητούνται άδειε. Η οικονομική στήριξη είναι κρισίμου σημασία, κυρίω σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Στρατηγικέ για ελαχιστοποίηση των φραγμών του, ώστε να χορηγούνται αυτέ οι άδειε στον τόπο εργασία. Σημαντικό. Προγράμμα την επιστροφή στην εργασία είναι σημαντικότατα. Διότι υπάρχει ο φόβο από του ανθρώπου ότι θα απομονωθούν από τον τόπο εργασία και ότι θα, θα επιστρέψουν δεν ξέρουν, θα έχουν την ίδια δουλειά. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και σε επίπεδο τόπου εργασίας οι πρακτικές των εργοδοτών επηρεάζουν άμεσα τις συμπεριφορές και την οτροπία των γονέων. Μπορώ να τα αναφέρω αυτό αργότερα. Σε αυτό εδώ το γράφημα φαίνεται να μην έχει σχέση με αυτά που συζητάμε, αλλά φαίνεται τι χρόνος ξοδεύεται στις διάφορες δραστηριότητε στην Ευρώπη και είναι για τον έλεγχο για τις συνθήκες εργασίας που κάναμε το 2010. Και βλέπετε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Από τη μία πλευρά οι άντρες ε, έχουν περισσότερες άδειες πληρωμένες, ε, που πληρώνονται. Δουλεύουν περισσότερο επί αμοιβή ε, από ότι οι γυναίκες. Οι γυναίκες όμως δουλεύουν πολύ περισσότερο προσέχοντας τα παιδιά από ότι οι άντρες. Οι άντρες μετά, κυρίως αυτοί που είναι ανάμεσα στα 35 και 49, στην ακμή της ηλικία τους και που έχουν παιδιά συνήθως, λένε ότι δεν ταιριάζει καλά ο χρόνος εργασίας με τις υποχρεώσεις εκτός ε, εργασίας συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών υποχρεώσεων. Η ισορροπία εργασίας οικογενειακής ζωής είναι κακή σύμφωνα με τους άντρες που είναι ηλικίε μεταξύ 35 και 49 και αυτό μας εξέπληξε. Λοιπόν, κλείνω. Ε, πρώτα απ' όλα, υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Είδα ότι οι άντρες θέλουν δείχνουν ότι ανησυχούν με την ισορροπία ιδιωτική ζωής και εργασία. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Ο επιμερισμός ε, της άνευ αμοιβής εργασίας είναι ανισόρροπος. Κάτι μπορεί να γίνει εκεί. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα κίνητρα, κυρίως τα οικονομικά κίνητρα ε, για αυτού του είδους τις άδειε. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τα νοικοκυριά έχουν το αναγκαίο εισόδημα για να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους η ένταξη όταν επιστρέφουν από τόπο εργασία. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι πάρα πολύ σοβαροί. Εκπροσωπούν του εργοζόμενου, του εργοδότε. Είναι στην καλύτερη δυνατή θέση να γνωρίζουν τι συμβαίνει στον τόπο, στον χώρο εργασία και πώ να εφαρμόσουν τι πολιτικέ. Άρα θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στι συζητήσει. Διοικητικοί, νομικοί, οικονομικοί περιορισμοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επίση. Αυτό είναι κάτι που συζητήθηκε επανειλημμένα εδώ οι περισσότερες εταιρείες μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν περιπλέξουμε την κατάσταση όσον αφορά ε, τα διοικητικά θέματα και τα νομικά θέματα θα είναι κάτι άχρηστο και θα πρέπει να συμμετάσχουν και οι άντρες στη συζήτηση. Η μητρότητα είναι σαν ταγκό, χρειάζονται δύο γι' αυτό. Οπότε οι πατεράδες συμμετέχουν, οι άντρες συμμετέχουν, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Κλείνοντας λοιπόν, οι πολιτικές πρέπει να είναι μεταμορφωτικές ούτε συμπίν. Δηλαδή η νέα νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αλλαγή της πραγματικότητας, την εξέλιξη και θα πρέπει να συζητούμε τα θέματα, να κάνουμε εκστρατείες λοιπά Αυτά είναι σημαντικά και να προχωρούμε σε πολιτικές που διαμορφώνουν μια διαφορετική κατάσταση. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Καμπρίτα. Σπουδαία δουλειά κάνατε με τις αναλύσεις της άδεια μητρότητας και πατρότητας στις 28 χώρες μέλη της Ένωσης και αυτό αποτελεί και τη στέρεα βάση για τη μελλοντική μας δουλειά. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μαρία Αρενά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ στην μελέτη αυτή που μας υποβάλλεται και μας δίνει πολλές πληροφορίες όσον αφορά τη σημερινή πραγματικότητα στις χώρες της Ευρώπης και μας βοηθά πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την παρουσίαση που έκανε. Όπως και εσείς κυρία Πρόεδρε αισθάνομαι πραγματικά παράξενα και κάπως προσβεβλημένοι, όπως και εσείς, δεδομένου ότι το θέμα μας είναι πολύ σημαντικό. Είναι τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη, η οποία διέχεται από μεγάλες δυσκολίες σήμερα. Και πολύ μικρή πρόεδρος έχει επιτευχθεί σε θέματα που αφορούν τη γυναίκα. Και το γεγονός ότι είναι από το Συμβούλιο σήμερα αποδεικνύει την έλλειψη ενδιαφέροντος για το θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σήμερα. Πρέπει λοιπόν να ομολογήσω ότι δεν, είμαι και πάρα, δεν με εκπλήσει και πάρα πολύ το θέμα αυτό, διότι όσον αφορά τη σχετική οδηγία είναι κάπως φαντασματικό το συμβούλιο. Εμείς δύσκολα μπορούμε να διαπραγματευτούμε κάποιον που είναι ένα φάντασμα, που δεν εμφανίζεται, που δεν έχει ολοκληρώσει την απόψή του και που δύσκολα μπορεί να συγκαλέσει σε ένα συμβούλιο ένα συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθούν τα θέματα αυτά που αφορούν τη γυναίκα. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ αποκριστάλλωστε στην προηγούμενη θητεία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε ευθύνες με τη θέση που εξέφρασε και σήμερα αναμένουμε, αναμένουμε το Συμβούλιο να ασχοληθεί εκ με το θέμα αυτό που αφορά τις γυναίκες την προστασία των γυναικών στον εργασιακό τους χώρο, των ε, γυναικών που πρέπει να προστατεύονται όταν είναι σε ενδιαφέρουσα στο χώρο της εργασίας σε σχέση με τις ε, ε, βαριά δύσκολη εργασία, την νυχτερινή εργασία, τα χημικά τοξικές ουσίες, την προστασία των γυναικών που έχουν ένα παιδί και είναι σε κατάσταση έμβιας το Συμβούλιο πραγματικά συνειδητοποιεί ότι σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες που βιώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις και απλώς και μόνο τι κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μας δείχνει τα νότα του και λέει ότι το θέμα αυτό δεν αξίζει καν να συζητηθεί σε ένα σχέδιο σημερινή διέκτηση ενό Συμβουλίου Θα πρέπει λοιπόν και εμεί να απομισθούμε τι ευθύνε, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επί του θέματο, να συνεχίσουμε ε, δεδομένου ότι αφορώνται οι γυναίκες να επιμένουμε για τα θέματα αυτά, αλλά αφορά και την ε, ε, γεννητικότητα στην Ευρώπη, τα ποσοστά τις οποίες συνεχίζουν να μειώνονται σημαντικά. Σήμερα στην Ευρώπη δεν αποφασίζει κανείς εν μία νυχτή να κάνει ένα παιδί. Το να φέρει στον κόσμο αυτό ένα παιδί είναι μία ευθύνη. Ευθύνη που μεταξύ άλλων ε, ενέχει το θέμα της προστασίας. Δεν αποφασίζει κανείς το έτσι να κάνει ένα παιδί. Αν λοιπόν εμείς που είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιες πολιτικές δεν μπούμε στα νέα ζευγάρια ότι τη μέρα που θα έχουν ένα νέο παιδί θα τα υποδεχθεί σωστά η κοινωνία στην οποία ζουν, δεν θα κάνουν παιδιά. Και οι νέες μητέρες τι πρέπει να διαλέξουν μεταξύ της οικονομικής τους αυτονομίας, δηλαδή τη δουλειά τους και τη μητρότητα. Και σήμερα επέλεξαν. Επέλεξαν να μην κάνουν παιδιά. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να έχουμε αύριο, διότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Αυτή την Ευρώπη φτιάχνουμε. Τα παιδιά που δεν θα κάνουμε σήμερα δεν θα τα έχουμε ούτε σε 10 χρόνια, ούτε σε 15 χρόνια, ούτε σε 20 χρόνια. Δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση με δημογραφικό έλλειμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό διεξοδικότητα. Και παρακαλούμε το θέμα αυτό το δημογραφικό, το σοβαρό, το συμβούλιο, το λάβει υπόψη και να ασχοληθεί. Επίση, σε σχέση με του στόχου στου οποίου ε, θέσαμε στα πλαίσια τη Ευρώπη του 2020, να απέχουμε από την υλοποίηση. Μπορούμε να πούμε από την πλευρά ότι όντω πρόκειται για διάκριση, το να μην μπορούμε να έχουμε ε, πολλές ε, γυναίκες στις θέσεις απασχόλησης τις σημερινές. Οι γυναίκες είναι ένα σημαντικό μέρος της ε, εργασιακής δύναμης. Μπορούμε σήμερα αυτή την σημαντική αναλογία στην αγορά εργασίας που είναι οι γυναίκες να τις χάσουμε. Οι γυναίκες είναι όλο και πιο μορφωμένες, έχουν όλο και περισσότερες γνώσεις, έχουν όλο και περισσότερα επαγγελματικά προσόντα και έτσι δεν χάνουμε μόνο τις γυναίκες αλλά και την ευφία τους. Και στην ευφία έχουμε κάνει μεγάλες επενδύσεις. Άρα μας κοστίζει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνουμε ως πολιτικοί. Δηλαδή κάνουμε μεγάλες επενδύσεις για την εκπαίδευση των γυναικών και χαίρομαι που γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά από την άλλη αυτές οι γυναίκες οι οποίες έχουν μορφωθεί δεν βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Είναι απαράδεκτη λοιπόν αυτή η κατάσταση. Αυτό το οποίο προτείνουμε λοιπόν και σε σχέση με αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα είναι να μπορέσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε μία οδηγία του 1992. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και όπως είπατε, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση αυτή, όσον αφορά το ποσοστό απασχόληση των γυναικών, τις άδειε μητρότητας, την, ε, ε, τα χρήματα, τις αμοιβέ, θα πρέπει να δούμε λοιπόν εμείς πώς σήμερα Εξετάζοντας όλα αυτά τα συστήματα, να δούμε ποιο λειτουργεί καλύτερα, πώς μπορεί ό,τι καλύτερο να είναι προσβάσιμο για όλες τις γυναίκες, ώστε να φτάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα υπάρχουν διακρίσεις κατά των γυναικών, διακρίσεις οι οποίες ε, είναι διακρίσεις που κρύβονται κατά κάποιο τρόπο, διότι όταν πάει κάποιο, κάποια γυναίκα μάλλον να εργαστεί, ο εργοδότη δεν σκέφτεται αν έχει τα ίδια προσόντα με έναν άντρα ή αν είναι ικανή να ασκήσει τα καθήκοντα τη θέση που τη ζητείτε. Το πρώτο που σκέφτεται είναι μήπω κάνει παιδιά και πάρει άδεια μητρότητας και φύγει για τη δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να τα επεξεργαστούμε για να προστατεύσουμε τι γυναίκε για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μία κάποια ισορροπία μεταξύ του επαγγελματικού άχθους και των οικογενειακών υποχρέωσεων για γυναίκα. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, όχι με φάντασμα όμως, μεταξύ ημών, αλλά και με ένα συμβούλιο που θα μας επιτρέψει να κάνουμε διαπρόμεση και να προχωρήσουμε. Διότι σήμερα έχουμε τα τρία θεσμικά όργανα, τα οποία θα πρέπει να σέβονται οι μεν τους δε και Καμή, κανένα από αυτά τα τρία θεσμικά όργανα δεν είναι ανώτερο από το άλλο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σήμερα πρέπει να πω ότι δεν γινόμαστε σεβαστοί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή το ίδιο δεν γίνεται σεβαστή. Δεδομένου ότι ένα από τα θεσμικά όργανα δεν ανέλαβε τι ευθύνε του. Ζητούμε λοιπόν από το Συμβούλιο να αναλάβει τι ευθύνε του, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και η οδηγία REFIT απειλεί ό,τι δουλειά έχει επιτελεστεί από τα άλλα δύο θεσμικά όργανα να χαθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι αν πάνε στον κάλαθο των αχρήστων ότι κάνουμε, θα πούμε τι είμαστε, πολιτικοί που ασχολούμαστε με άχρηστα πράγματα. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Και τι θα πει η Κομισιό. Εμείς είμαστε ε, υπάλληλοι που δουλεύουν για χρηστά πράγματα. Αυτό έμεσα μας λέει το Συμβούλιο. Υπάρχουν όμως πολίτες που δεν θέλει κανείς να τους θεωρεί άχρηστους ή ελάσσονος σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Εάν δεν κάνουμε κάτι για το θα χάσουμε πέντε χρόνια παραπάνω. Δηλαδή, θα έχουμε στην Ευρώπη την οδηγία του 1992, η οποία όμως Ενδεχομένω θα τροποποιηθεί κατά κάποιο τρόπο αν όλα πάνε καλά το 2025. Δεν είναι αποτελεσματικό τρόπο εργασία των θεσμικών οργάνων αυτό. και δεν εκπλήσωμε που πολλέ φορέ βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ αυτών που πίστευαν οι πολίτες όταν προσχώρησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτού που συμβαίνει σήμερα και τα δικά του συναισθήματα. Θα ήθελα λοιπόν ο καθένας να υποφεληθεί τη ευθύνη του Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Ρενά. Σας δείχνει και το χειροκρότημα πώς εκτιμούν οι συνάδελφοί μου το γεγονός ότι σκέφτεστε να εργαστείτε με τον τρόπο που εξηγήσατε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τεσούσης, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διευθύντρια δηλαδή, της Γενικής Διεύθυνσης Καταναλωτών και Δημόσιας Υγείας. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μετά από τέτοιο πάθος που ε, έδειξε με την ομιλία της η κυρία Αρένα, ακόμα και αν εγώ θεωρώ ότι έχω και εγώ πάθος, βεβαίω δεν μπορώ να σας συναγωνιστώ, κυρία Αρένα. Ωστόσο, έχω έρθει ενώπιόν σας για να συζητήσουμε αυτή τη σημαντική πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άδεια μητρότητας. Μια από τις οδηγίες που έχουμε στη Γενική μας Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών υπό την ευθύνη της ε, Επιτρόπου κ. Γιούροβα. Mm. Μέρος του χαρτοφυλακίου της κ. Γιούροβα βεβαίως είναι και αυτό. Όπως πολλές εξημών Απογοητεύτηκα κι εγώ που οι συνομοθέτες δεν μπόρεσαν ακόμη να βρουν κοινό έδαφος για την πρόταση αυτή. Και όχι μόνον επειδή εμείς είμαστε δημόσια αξιωματούχοι και κάνουμε τελικά τη δουλειά μας όπως θεωρούμε πιο ενδεδειγμένο, αλλά και διότι πιστεύαμε και νομίζω ότι πιστεύαμε αυτό που προτείναμε όταν προτείνουμε κάτι, οφείλουμε να αιτιολογήσουμε γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει σχετική ρύθμιση. Για μας πάντοτε η πρόταση ήταν καλή και καλά ισορροπημένη. Επειδή είμαι και μητέρα και έχω ένα παιδί, μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο στον κόσμο. Για τη γυναίκα, αλλά όχι μόνο για τη γυναίκα. Μίλησε η κυρία Ρενά για ευθύνη. Η ευθύνη δεν αναλαμβάνεται ούτε πρέπει να αναλαμβάνεται μόνο από τη μητέρα. Το μέγα βάρος δεν είναι βαρύ το βάρος αυτό, αλλά αν δείτε τέλος πάντων ολόκληρη τη ζωή μιας γυναίκας θα δείτε ότι είναι μεγάλο το βάρος που ε, καλείται να σηκώσει. Αυτό λοιπόν το βάρος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλες και όλοι και άντρες και γυναίκες είμαστε υπεύθυνοι για να βρούμε λύσεις. Καθώς ο χρόνος περνά και έχει κατατεθεί η πρότασή μας, όσο περισσότερο περνά ο χρόνος, τόσο λιγοστεύουν οι δυνατότητες ε, έγκρισης. Είμαστε παγιδευμένοι τόσο καιρό σε μια κατάσταση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αποσύρει την πρόταση για να ξαναγίνει η προσπάθεια από την αρχή. Εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερα τις σοβαρές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την Ευρωβουλή και ιδιωτικότερα από εσάς κυρία Ρενά ως νέα εισηγήτρια ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιθυμώ να σας δηλώσω ότι σας στηρίζουμε για να μπορέσετε να βρείτε τη σωστή λύση για να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της γενική Διεύθυνσης, δηλαδή στο ύψιστο επίπεδο. Ε. Αλλά θα χρειαστεί την υποστήριξη όλων, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο περιμένει από το Κοινοβούλιο. Περιμένει το Κοινοβούλιο να μαλακώσει τις θέσεις του. Και ιδίως ό,τι αφορά την πλήρη εξίσωση των αμοιβών για όλη την περίοδο της ε, άδειας μητρότητας. Ξέρω ότι έχετε ήδη μια εναλλακτική πρόταση, αλλά αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει τώρα είναι να δοθεί μια πιο επίσημη μορφή σε αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύω τόσο πολύ στα τυπικά, προσωπικά όμως. Ε. Αν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε σωστά, χρειαζόμαστε κανόνες και χρειάζονται βέβαια και κάποια στοιχεία τυπικά. Όσοι γνωρίζετε, χρειάζονται δυο για να χορεύσουν ταγκό. Και ο άλλος ο σα σας είναι το Συμβούλιο και πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο του. Άρα, η Λεκτονική Προεδρία πρέπει να αποφασίσει πια πώς θα προχωρήσει. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι η Κομισιόν και εγώ προσωπικά και οι υπηρεσίες μου συζητούμε με την Προεδρία για να βρούμε και εναλλακτικέ δυνατότητες να προχωρήσουμε. Να καταστήσω ωστόσο κάτι σαφέ από τη σκοπιά της Κομισιόν. Ακόμα και αν ισχύσει το χειρότερο ενδεχόμενο και αποσυρθεί εντελώς η τρέχουσα πρόταση, δεν μπορούμε, ούτε θα εγκαταλείψουμε ποτέ τι γυναίκες. Ασφαλώς, δεν θα εγκαταλείψουμε δε τις μητέρες. Θα χρειαστεί να δούμε με μια φρέσκια ματιά το θέμα η Επίτροπος κυρία Γιούροβα ήδη το ανακοίνωσε αυτό, αλλά βέβαια μένει να δούμε πώς και τι ακριβώς θα κάνουμε, εάν η παρούσα απόπειρα δεν αποδώσει καρπούς τους επόμενους μήνες. Σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι οικογένειες βέβαια για να ξεσορροπήσουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή. Μίλησατε και για τις δημογραφικές αλλαγές. Με ε, μεγάλο ενδιαφέρον δεν παρακολουθώ την ανάπτυξη των απόψεών σας για το θέμα αυτό και θα παρακολουθήσω. Πολλές γυναίκες θέλουν να κάνουν παιδιά. Βέβαια και χρειαζόμαστε και πρέπει να δουλέψουμε και να αναπτύξουμε μια σταδιοδρομία. Είπατε ήδη κυρία Αρενά ότι, και βέβαια υπάρχουν και σχετικές στατιστικές, ότι οι γυναίκες έχουν, διαθέτουν πλέον υψηλότερα προσόντα από ό,τι στο παρελθόν. Όπως πάμε όμως, χάνονται τα ταλέντα αυτά, χάνεται και αυτό το σύνολο ταλέντων και μάλιστα σε μια εποχή όπου μειώνεται ο πληθυσμό αυξάνεται δηλαδή ο παγκόσμιο ταγωνισμό. Άρα, χρειάζεται να βρούμε μια στοχευμένη προσέγγιση για να εξασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα στο επάγγελμα και στην οικογενειακή ζωή για να επιτρέψουμε σε γυναίκες με παιδιά και να μπουν στην αγορά εργασία και να παραμείνουν. Βέβαια δεν είναι μονάχα να βοηθήσουμε τις γυναίκες, οπότε τις γυναίκες βοηθούν και τις οικογένειες. Αυτό πάλι θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε μία από τις ρίζες ε, του χάσματος στην αμοιβή, δηλαδή αμοιβή μεταξύ φίλων αλλά και στι συντάξει. Και να μοιραστούν βέβαια τι ευθύνε και για την οικογενειακή ζωή άνδρες και γυναίκες. Και δεν μιλούμε βέβαια μονάχα για τις γυναίκες όταν αποκτούν παιδιά. Μιλούμε και για τις γυναίκες σε κάθε πτυχή της ζωής. Και όταν έχουν παιδιά και όταν τα παιδιά ρωσταίνουν και όταν τα παιδιά και όταν οι γυναίκε φροντίζουν του γονεί και ούτω καθεξή. Δηλαδή, μιλάμε για όλη τη ζωή τη γυναίκα. Εγώ πια είμαι πεπισμένη ότι μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματο και ε, ζωής θα επιτρέψει και στις, και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προσελκύσουν επαγγελματίες μέσα σε αυτή τη, δηλαδή με σωστά προσόντα μέσα σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά. Και επιπροσθέτως, πολλές εργαζόμενες μητέρες υποπασχολούνται σε δουλειές που είναι χαμηλότερες από τα προσόντα που διαθέτουν λόγω έλλειψης ευκαιριών. Χρειάζεται λοιπόν να τις διευκολύνουμε να βρουν καλές δουλειές και μάλιστα να φτάσουν και μέχρι το επίπεδο του management. Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών την αγορά εργασίας θα έχει ασφαλώς θετική απήχηση και στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη και στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει ένα μείγμα πολιτικής συμφιλίωσης για να βοηθήσει τους γονείς που έχουν ανάγκη να εργαστούν. Μέτρα που πρέπει βέβαια να προσαρμοστούν στις διάφορες φάσεις της ζωής όταν τα παιδιά είναι πολύ νέα στην ηλικία, όταν θα αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο ή όταν άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα χρειάζεται να τα φροντίσουν. Πρέπει λοιπόν να καταργήσουμε τους φραγμούς στην οικονομική συμμετοχή των γυναικών, συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία. Να προωθήσουμε την κοινή ανάληψη των οικογενειακών ευθυνών και εν τέλει αξιότιμες ευρωβουλευτές έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Όπως είπα ήδη, κατ' επανάληψη μάλιστα και στις συναδέλφους μου, πρόκειται για μακροπρόθεσμο έργο. Με μεγάλη χαρά θα ακούσω τις απόψεις σας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις σημαντικές προκλήσεις σήμερα. Να συνεχίσουμε δηλαδή τον αγώνα για να προωθήσουμε μια ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έτσι ώστε περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας και περισσότεροι άνδρες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνεται πλέον να μείνουν στο σπίτι να φροντίσουν τις οικογένειες και τα παιδιά. Αξιότιμες ευρωβουλευτές, η Κομισιόν θα είναι πάντα στο πλευρό σας για να δουλέψει μαζί σας, για να βρεθούν οι σωστές λύσεις για μια ισορροπία μεταξύ ε, δουλειάς και ζωής. Αυτό που εν τέλει θέλω να σας πω είναι ότι εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα δω το ρόλο της γυναίκας ως ρόλο θύματος. Οι γυναίκες έχουν προσόντα. Οι γυναίκες έχουν μάλιστα τρομερά προσόντα σήμερα. Είναι overqualified και βεβαίω έχουν και δικαιώματα. Και άντρες έχουν δικαιώματα. Δεν λέω. Και δεν ξέρουν και τι χάνουν όταν δεν είναι κοντά στα μικρά παιδάκια τους. Αν όμως δουλέψουν άντρες και γυναίκες μαζί θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. E, e, Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Γενική Διευθύντρια, mm. κυρία Μίχου. Ας αρχίσουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτα, οι σκληρές της από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. κυρία Ζαβόρσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για τη μελέτη που παρουσίασε ο εξαίρετος εμπειρογνώμων και που μας πρόσφερε και μια εικόνα της καταστάσεως, πώς διαμορφώνεται δηλαδή στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της εγώ είμαι Σλοβάκη, ή Σλοβάκα. Έχουμε 34 εβδομάδες υποχρεωτική άδεια μητρότητας. Όμως, αυτό δεν είναι ακριβές, όπως το περιγράψε ο εξαίρετος εμπειρογνώμων. 34 εβδομάδες ισχύουν για γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες τους. Έχουμε βέβαια και δυνατότητα μάλλον για αυτές τις τελευταίες γυναίκες, δηλαδή που μεγαλώνουν τα παιδιά μόνες τους, έχουν ε, τη δυνατότητα να πάρουν μακρότερη άδεια μητρότητας. Τώρα, εκφράζω τη λύπη μου που δεν είναι παρούσα εκπροσώπηση του Συμβουλίου. Γίνεται σήμερα άλλη μια συζήτηση βέβαια εδώ για ε, το θέμα αυτό και από όσο θυμόμαι ποτέ το Συμβούλιο δεν ήταν παρόν ούτε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν θυμάμαι ούτε μία φορά που να ήταν παρόν το Συμβούλιο σε τέτοιες συζητήσεις που έχουμε διεξαγάγει εδώ. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν ήταν ενωμένο στην ψηφοφορία. Εγώ πάντως ψήφισα υπέρ της εκθέσεως της κυρίας Εστρέλα τότε αν και όχι όλοι οι συναδελφοί μου έπραξαν το ίδιο, χαίρομαι που η κυρία εισηγήτρια, η κυρία Αρενά, κάνει αυτή την πρόταση, έκανε ήδη δηλαδή την πρόταση αυτή, που τη βρίσκω πολύ επικοδομητική. Όλες οι συζητήσεις που έχουν διεξαχθεί έως τώρα, δείχνουν ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών εμένει στις θέσεις της. Βέβαια θα προχωρήσουμε καλύτερα εάν συμπαραταχθούν με την γενναιόδορη αυτή πρόταση της κυρίας Αρενά περισσότεροι ευρωβουλευτές. Πρέπει να συνομιλήσουμε και με το Συμβούλιο. Εγώ πάντως εξ ονόματος της κοινοβουλευτικής μου ομάδος τάσσομαι υπέρ της δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας στο επίπεδο του Συμβουλίου που να αντιδράσει, να παρουσιάσει τη θέση του Συμβουλίου απέναντι στην πρότασή μας. Δεν γνωρίζουμε βέβαια ποια μπορεί να είναι αυτή η θέση του Συμβουλίου. Πάντως, να μην δυσμονούμε ότι στην οδηγία για την οποία μιλούμε Πρόκειται για την προστασία των γυναικών, των γυναικών που θυλάζουν Αυτό δε είναι το περιεχόμενο που είχε κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλώνουμε έτοιμες να συζητήσουμε το Συμβούλιο ανα πάσα στιγμή είμαστε διατεθειμένες και να προχωρήσουμε σε συμβιβασμούς. Εάν γίνει δυνατό να διεξαχθεί η συζήτηση με το Συμβουλίο, τότε θα μπορέσουν να προσεγγίσουν και οι θέσεις μας. Και θα έχουμε βέβαια τότε καλύτερες προϋποθέσεις για να προωθήσουμε την λύση. Η κυρία Γενική Διευθύντρια, αλλά και η κυρία Εισηγήτρια, μίλησαν και εξήγησαν τη θέση των γυναικών. Εξήγησαν επίσης ποια είναι η δημογραφική κατάσταση των κοινωνιών μας. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των σοβαρών αυτών προβλημάτων, πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο τολμηρά. Δεν νομίζω ότι η παρούσα οδηγία θα αποτελέσει τη λύση του δημογραφικού προβλήματος. Παρ' όλα αυτά θα βελτιώσει σημαντικά την θέση των ε, εγγύων και των γαλουχουσών γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Οκτώ συνάδελφοι έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Έκλεισε ο κατάλογος. Δύο λεπτά ο καθένας, αν έχετε την καλώση. Η κυρία Μπέλντερ από την ομάδα της Άλτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρους της Μπέατριξ Μπεκέρα που είναι σκιώδης της Άλτε και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα. Προσθέτω και εγώ τις ευχαριστίες μου όσον αφορά την παρουσίαση που την βρήκα επικοδομητική ε, και ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ και την κυρία Ρίνα για τη σκληρή δουλειά που έκανε προσπαθώντας να βρει μια διέξοδο. το έργο, το έργο της το εκτιμούμε και βρήκε έναν τρόπο να στείλει σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Δηλαδή το Κοινοβούλιο έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες. Το μπαλάκι τώρα είναι στο γήπεδο του Συμβουλίου και ρόλος του είναι να κινηθεί επικοδομητικά και υπεύθυνα. Όμως είναι απαράδεκτο μια οδηγία να αποσύρεται βάση μη συμμετοχή του Συμβουλίου. Και εμεί είμαστε πολύ απογοητευμένοι, όπως όλοι οι άλλοι, διότι η Λετωνική Προεδρία επέλεξε να μην παρίσταται εδώ για να συμμετάσχει στη συζήτηση. Η μέθοδος που περιέγραψε ο πρόεδρος Γιούνκερ, δηλαδή ότι θα αποσυρθεί η οδηγία αν το Συμβούλιο δεν συμμετάσχει, στις συζητήσει, και στι εργασίε δημιουργεί ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για όλου μα. Πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού. Υποχωρεί η ισότητα. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο ήταν να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε την κυρία Γιουρόβα και την εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκληρή του δουλειά. Ε, ξέρουμε ότι μα στηρίζετε και σα ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Συμβούλιο να ξεφύγει. Ευχαριστούμε κυρία Αρίνα, θα συνεργαστούμε μαζί σας ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να ξεφύγουμε το τέλμα. Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ευρώπης ε, ζητούν από εμά να το προθίσουμε το θέμα. Δεν είναι αποδεκτό να έχουμε στα χέρια μας πρόταση του 1992 που θα είναι το μόνο που θα μας μείνει στα χέρια μας αν τελικά καταπέσει η παρούσα πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ορτασούν. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω απόλυτα με την συνάδελφο Μάρια Ρένα σε σχέση με την οδηγία αυτή. Νομίζω ότι όλο και περισσότερη αγανάκτηση υπάρχει. Το ξέρει η Κομισιό. Δεν είναι το Συμβούλιο. Γράφει ότι όλοι πιστεύουν ότι θα ψηφιστεί η οδηγία αυτή. Και θα επιδεινωθούν οι ανισότητες και αν δεν προχωρήσουμε στην αναγνώριση κάποιων δικαιωμάτων θα είναι χειρότερα τα πράγματα και οι ανισότητες. Και η οικονομική κρίση δεν είναι μία δικαιολογία για να δημιουργήσει κανείς τροχοπέδι σε τέτοιου είδους οδηγίες, τέτοια θέματα. Ξέρουμε ότι όταν έγινε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν εκ μέρους κάποιων πάρα πολλές ε, ε, διακηρύξεις λέγοντας ότι εφόσον έχουμε οικονομική κρίση δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ισότητα. Αυτό είναι ένα ε, κριτήριο πολιτικό που επικαλέστηκαν πολύ όχι μόνο για το θέμα αυτό αλλά και για πολλά άλλα. Τώρα, ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Επιτροπής και κατανοώ ότι προσπαθείτε εσείς να κάνετε ό,τι μπορείτε για να ξεμπλοκαριστεί το όλο θέμα του φάκελος. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε και πόσο συνεισφέρετε. Δηλαδή, πήγε στη ρηφή το φάκελος. Τι, ποιο άρθρο της συνθήκης σας επιτρέψει να το κάνετε αυτό. Το 2.94 που λέει ότι μετά την πρώτη ανάγνωση πρέπει να μας επιτρέψει, επιτρέψει ο Συμβούλιο την έκθεση ή το 2.92, δηλαδή για κάτι που θα διευκολύνει διαπραγματεύση. Δεν γίνεται τίποτα όμως. Όλα πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω το εξή λοιπόν. έχει το, την υποχρέωση το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο να στείλει την της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς είμαστε στην λογική της διαπραγμάτευσης. Είτε πρώτη είτε δεύτερη ανάγνωση. Θα πρέπει να μας κάνει μία πρόταση στο Συμβούλιο και θα μιλήσουμε για ό,τι λείπει και χρειάζεται για τις ημέρες, για τις άλλες, για τη Μητρόπιτα, για την ε, αντισταθμίσματα, για τις αμοιβέ. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό. Δεν μπορεί να μας λέει κάτι το Συμβούλιο χωρίς να μας στέλνει την, ε, ε, το κείμενο της διαπραγμάτευσης. Έχω την εντύπωση ότι όλοι θέλουν να προχωρήσει αυτός ο φάκελος. Και αν δείτε κι εσείς και κατανοήσετε ότι αυτή είναι η σημαντική στάση που πρέπει να κρατήσετε, παρακαλώ να λάβετε τις ευθύνες σας. Μην στείλετε τα πράγματα στο κάλαθο των αχρήστων. Προχωρήστε το. Και βεβαίω, η ιδέα που τέθηκε εδώ, να δημιουργηθεί μία ομάδα εργασία για να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε, με βρίσκει σύμφωνο ότι είναι εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκέρκ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Να δούμε αν θα καταφέρω. Θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση. Θα μιλήσω γερμανικά κατά τα υπόλοιπα. Μου φαίνεται δε εκπληκτικό ότι ορισμένοι δουλεύουν εδώ και μια δεκαετία για την οικογενειακή πολιτική και εξακολουθούν να έχουν τη λάθος προσέγγιση. Και στη μελέτη είδαμε σύγκριση μεταξύ πατέρα και μητέρας. Εσείς κύριε αναλυτά, ήσασταν ποτέ έγκυος, μεγαλώσατε κανένα παιδί. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά. Και βέβαια δεν έχω ζήσει καμιά εγκυμοσύνη. Ούτε και θύλασα παιδί. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Δεν είναι άδεια. Στα γερμανικά λέμε Urlaub. Άδεια δηλαδή μητρότητας. Δεν είναι άδεια. Είναι δουλειά σκληρή. Το να μιλάμε εδώ τώρα για άδεια μου φαίνεται ήδη ότι δυσφημίζει την έννοια. Τα παιδιά μπαίνουν στην κοινωνία. Τα παιδιά τα φτιάχνουν οι γονείς για να εξασφαλίσουν στο μέλλον τις συντάξεις άλλων. Αυτό που δεν βλέπω εδώ είναι μια σύγκριση μεταξύ γονιών και άτεκνων. Αυτή τη σύγκριση χρειαζόμαστε. Όχι φτωχούς και πλούσιους γονείς. Χρειάζεται μια αντιπαράθεση, νομική αντιπαράθεση, ε, ανάμεσα σε γονείς και σε άτεκνους. Αυτό είναι το σημαντικό όσους νόμους και να φτιάξετε, πάντα θα υπάρχει μια αρνητική διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γονιών. Η οικογενειακή πολιτική που ασκείται στην Γερμανία εδώ και 50 χρόνια, και βέβαια σε ένα μέρος της Γερμανίας μόνο 20 χρόνια, έχει αυτό το σφάλμα. Τα παιδιά αποτελούν ένα βαρύ καθήκον. Να μην μιλούμε για δικαιώματα των γυναικών και δικαιώματα των ανδρών είναι σωστό αυτό βεβαίω και πολύ καλά κάνετε εδώ και τα συζητάτε. Αλλά θα έπρεπε μάλλον να βάλουμε, να αντιπαραθέσουμε νομικά, όπως είπα, γονεί και ατέκνους. Τότε να μιλήσουμε όχι μόνο για το κοινωνικό βάρος που σημαίνει το παιδί, αλλά και την ευθύνη για το μέλλον της κοινωνίας μας. Πού είναι αυτοί που φέρουν κυρίως οι γονείς. Ευχαριστώ κύριε Ζούμπερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αυτούς που φερουν κυριω οι γονεις ευχαριστω μέχρι τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα που τίθεται εδώ. Εξαρτάται πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει εδώ και στο Συμβούλιο και στις συζητήσεις όλοι είναι υπέρ συμφωνιών στα οικονομικά είναι υπέρ των περικοπών, κοινωνικών περικοπών, οικονομικών περικοπών κλπ. Όπως γίνεται συζητήσει και στο Eurogroup. Αυτή η προσέγγιση όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς. Ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το εξή. Το ζήτημα που συζητούμε για εκείνους που δεν θέλουν να το δουν σαν θέμα δικαιωμάτων, ανθρωπιάς μπορεί να οδηγήσει και σε οικονομική προσέγγιση, άμα θέλετε, να λύσουμε έτσι τα πράγματα. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό τεράστιο. Και η αύξηση των δικαιωμάτων για την άδεια μητρότητας και πατρότητας ε, θα έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Ποια είναι η αλήθεια. Αν δεν αλλάξουμε την κατάσταση σχέση με σήμερα, και η οικονομική κατάσταση θα περιπλοκεί ε, περαιτέρω. Λοιπόν, δεν πρέπει να μιλάμε για μητρότητα και πατρότητα σαν ατομικά δικαιώματα, αλλά έχοντας υπόψη και την κοινωνική κατάσταση των γονέων όταν έχουν ένα παιδί. Εκτελούν ένα κοινωνικό λειτουργήμα έναντι της κοινωνίας που θα πρέπει να στηρίζεται από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά τη χώρα μου, αν αληθεύει ότι σε κάποιες χώρες το ότι δεν υπάρχουν νομοθεσίες για να προστατεύουν εξίσου την πατρότητα για να μπορούν οι γυναίκες να μένουν στο σπίτι όταν δεν είναι σωστή νομοθεσία τελικά πέντε το αποτέλεσμα δεν κάνουν παιδιά οι γυναίκες δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα στο σπίτι. Διότι ε, δεν τα καταφέρνουν οι οικογένειες να τα φέρουν βόλτα με έναν μόνο γονιό να εργάζεται. Είναι αδύνατο να επιβιώσουν. Και το αποτέλεσμα είναι να αποφασίσουν τα, να μην κάνουν παιδιά τα ζευγάρια. Πολλοί λένε θα κάνω παιδί αν μπορώ να το συντηρήσω. Αυτό δείχνει μια κάποια οριμότητα. Σχετίζεται κατά πολύ με τις κοινωνίες μας αυτή την εποχή. Όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου, θα ήταν καλό να ξέρουμε ποιες χώρες θέτουν εμπόδια. Οι κυβερνήσεις που το κάνουν θα πρέπει να επομιστούν τις ευθύνες τους. Και εμείς έχουμε ένα ρόλο να δείξουμε αυτή την ευθύνη. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να ξεκινήσει να βγάλει αυτό το θέμα από το κατάλογο των refit, να σκίσει και ίσως τελικά να βοηθήσει το Ευρωκοινοβούλιο σε διαπραγματεύσεις που ενδεχομένω να γίνουν με το Συμβούλιο. Αν ασκηθούν πιέσεις σε όλους τους τομείς, ε, θα είναι δυνατόν να το συζητήσουμε το θέμα. Ε, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Το Κοινοβούλιο πάντα ήταν ε, διαθέσιμο να συζητήσει η κυρία Εντίθε Στρέλα στην προηγούμενη θητεία έκανε ό,τι μπορούσε για να ζητήσει από το Συμβούλιο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο ποτέ δεν υπαναχώρησε, ποτέ δεν είπε ότι είμαστε διαθέσιμοι να μιλήσουμε αντιθέτως, μάλιστα. Αν υπάρχει εμπόδιο, ποτέ το εμπόδιο αυτό δεν δημιουργήθηκε από το Κοινοβούλιο παρά μόνο από το Συμβούλιο και μόνο. Κυρία Γιούτα, ευχαριστώ. Αισθάνομαι να συμμετέχω σε πρώτο πρόσωπο σε αυτό το θέμα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνο που θέλω να πω και πιστεύω ότι κάπου χάνεται από τη συζήτηση είναι αυτά που άκουσα από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρθηκε στο, την όλη προβληματική, το μεγάλωμα των παιδιών, την προβληματική του μεγαλώματος των παιδιών, σχέση άντρας, γυναίκας, εντός της οικογένειας για το μεγάλωμα των παιδιών. Δεν είναι αυτός ο πυρήνας του θέματος. Ο πυρήνας είναι αυτός. Να εργάζεται κανείς και να είναι έγκυος, να έχει κανείς την εγγύηση ότι θα ξαναβρει τη θέση εργασία της και να έχει τη δυνατότητα να κάνει τα παιδιά. Εγώ είμαι προνομιούχα, μπορώ να έρχομαι να δουλεύω τελευταία μέρα αλλά είμαι προνομιούχα. Δεν είμαστε όλες προνομιούχες. Πόσες Ευρωπαίες γυναίκες μπορούν να πάνε, πρέπει να πάνε εργαστούν διότι δεν έχουν την εγγύηση ότι θα έχουν οικονομική στήριξη ούτε μετά όταν ξαναβρούν τη θέση εργασίας τους. Είναι οι γυναίκες έχουν κουραστεί να περιμένουν οι γυναίκες πολίτες. Ήδη σε κάποιες χώρες υπάρχουν τα δικαιώματα. Χρειάζεται μια διεύρυνση, μια επέκταση. Από τη μελέτη φαίνεται ότι η χώρα μου είναι μία από εκείνες τις χώρες που έχει μεγαλύτερη άδεια ε, που χορηγείται. Υπάρχουν όμως πολλές σκιώδεις περιοχές και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες ε, που δεν μπαίνουν στατιστικά. Γυναίκες που δεν έχουν δικαιώματα ίσως διότι εργάζονται με σύμβαση και έχουν πολλά προβλήματα. Πρέπει αυτές οι κατεπίγουσες περιπτώσεις να μην αναβάλλονται θα πρέπει απόλυτα να μην αφήσουμε να καταπέσει αυτή η έκθεση, να μην εξαφανιστεί. Λυπήθηκα που άκουσα αυτά που μας είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεώρησε σαν να ήταν ήδη κάτι χαμένο, χαμένο παιχνίδι. Να θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται να απορριφθεί, να αποσυρθεί. Τώρα, το να θέσουμε έξι μήνες ε, σαν όριο είναι ελάχιστο. Ζητούμε πάνω απ' όλα να μην αποσυρθεί, να δοθεί χρόνος να προσπαθήσουμε να σπρώξουμε το θέμα ώστε τελικά και το Συμβούλιο να μην συμπεριφέρεται όπω κάνει, με την πλήρη απουσία του. Άρα είναι ανέφικτο να υπάρξει ένα διάλογο μαζί του. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι δεν μπορώ να μιλήσω στα ουγγρικά, διότι δεν υπάρχει διερμηνία. Θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά. Εξακολουθώ να πιστεύω στο παλιό ρητό του κινήματος των γυναικών. Ότι το προσωπικό είναι πολιτικό, χρησιμοποιώ το δίλεπτό μου, περίπου, για να μοιραστώ μια προσωπική ιστορία. Εμείς όταν παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις πολιτικοί, θα πρέπει να ακούμε πολλές προσωπικές ιστορίες πραγματικών γυναικών. Πάμε πίσω λοιπόν στο 92. Είμαι 28. Το πρώτο μου παιδί γεννιέται. Ζητώ δουλειά στο Συμβούλιο της Ευρώπης που μόλις είχαμε, είχε μπει η Ουγγαρία σαν προεκομιστική χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και κάνω αίτηση για δουλειά. Για νομικός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πήγα στη συνέντευξη, ε, έδειξα αποτελέσματα ιατρικής εξέτασης, ε, θέλαν να δούνε αν ιατρικά μπορούσα να εργαστώ, ε, να μου κάνουν ιατρικές εξετάσεις, έπρεπε να αγβηθώ και ένας μεσήλικας αρχίζει λοιπόν να χρησιμοποιεί το στιθοσκόπιό του στο στήθος μου. Ξαφνικά με κοιτάει συνοφριωμένος, καχύποπτος και με ρωτάει θυλάζεται ανοίγει το φάκελό μου και λέει το παιδί σας είναι εννέα μηνών και εξακολουθείτε να τον θυλάζετε. Η δίκευσή μου ήταν ποινικό δίκαιο και αμέσως σκέφτηκα αυτά που βλέπεις σε, σε ταινίε, την προειδοποίηση που σου κάνουν. Προσέξτε τι θα πείτε, μπορεί να ληφθεί η υπόψη σας εναντίον σας. Και θεώρησα μήπως αυτό είναι έγκλημα στη χώρα. Τι είναι, ποινικό αδίκημα, τι είναι. Είμαι δεινόσαυρος που ζω σε λάθος εποχή. Ήμουνα σίγουρη ότι έκανα κάτι πάρα πολύ κακό. Του λέω, ναι, ναι, το κάνω. Ίσως ε, έχω ελαφρυντικά, το παραδέχομαι, ε, αλλά το κάνω. Ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, απογοητεύτηκε. Μου λέει, εννιά μηνών παιδί και το φυλάζεται. Δεν κάνει καλό στο παιδί, και είναι άχρηστο για το παιδί, είναι απαιτητικό για το σώμα σας και είναι εμπόδιο για σας να εκτελέσετε σωστά τα καθήκοντά σας. Σας δίνω αυτό το φάρμακο, αλήθεια σας λέω, δεν είναι φίβρα τώρα, πάρτε αυτό το φάρμακο, πάρτε την τάδε δόση και θα στερέψει το γάλα σας. Και σαν γιατρός σας το συστήνω αυτό. Δεν θα λησμονήσω ποτέ πώς αισθάνθηκα, πόνο, ταπείνωση, μοναξιά. Επέστρεψα στο ξενοδοχείο. Και κάθε φορά που είμαι στο Στρασβούργο, δεν ξέρω, πήγα στην Πλάσ Κλεμπέρ. Υπάρχει ένα μικρό ξενοδοχείο. Με βλέπω τώρα, σαν να είναι τώρα, 24 χρόνια πριν. Κάθομαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου, με τα χάπια στο χέρι και αισθάνθηκα ότι έκανα φρικτό λάθος που μοιράστηκα μια... Μάλλον είπα και σε κάποιον άλλον που είχε κάνει αίτημα για δουλειά, έναν Ούγγρο που ήταν ψυχολόγος και δικηγόρος από την Ουγγαρία. Και μου λέει αυτός, σαν ψυχολόγος, ναι συγγνώμη ακρηγόρησα, όλο λέω ιστορίες για γυναίκες, αλλά είναι Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών βλέπετε. Ποιο είναι το τέλος της ιστορίας. Ήταν ψυχολόγος αυτός, με συμβούλεψε να πάρω τα χάπια και να σταματήσω να θυλάζω. Δεν το έκανα και αυτό είναι το καλό τη ιστορία. Αποφάσισα να μην το κάνω. Συνέχισα να θυλάζω για άλλου τρει μήνε και γέννησα κι άλλα δύο παιδιά. Αλλά ταυτίζομαι με τι γυναίκε που εξακολουθούν να αισθάνονται μοναξιά, ότι πονούν, ότι είναι ταπεινωμένε και έχει χρειά φίλου. Λυπούμε. Λοιπόν, σα σέβομαι που λέτε ότι δεν πρέπει να, να δίνουμε απόχρωση φίλου στο θέμα ότι δεν πειράζει αν οι γυναίκες. Στην πραγματική ζωή δεν αισθάνεται κανείς τόσο ταπεινωμένος. Όλοι χαίρονται τη συμμετοχή του πατέρα. Έχουμε άλλα τρία θέματα στην μερίσια διάταξη, λέει Παρακαλώ, συντομεύετε. Ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε ακουράσεις πραγματικές γυναίκες, να λένε τις πραγματικές τους ιστορίες για το πώς η μητρότητα, ο θυλασμός, η εγκυμοσύνη και η γένα επηρεάζουν την εργατική του ζωή. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madame Petir, please. Ευχαριστώ κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό το θέμα. Λυπάμαι που δεν είναι εδώ εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Να πω στην Επιτροπή ότι την περασμένη εβδομάδα μαζί με την Πρόεδρο και άλλο συνάδελφο επεσκέφθημεν τη Λετωνική Προεδρία σαν αποστολή τη Επιτροπής Γυναικών. Συζητήσαμε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεω και συμπεριλάβαμε το θέμα στο πρόγραμμά μας. Ζήτησα εκ μέρου Επιτροπής μας από το Συμβούλιο να προβάλλει τη θέση του και να μας ενημερώσει πότε προτίθεται να το συζητήσει, να συζητήσει την οδηγία λάβαμε μια άκρος παράδοξη απάντηση και αόριστη όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Το Συμβούλιο συνέστησε το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει επιθέσεως επί της οδηγίας και μετά να δει το Συμβούλιο τι θα κάνει. Θα ήθελα να τονίσω ότι χρειαζόμαστε καλή νομοθεσία, καλούς κανονισμούς για να προστατεύουμε τις μητέρες και να δίνουμε τη δυνατότητα στις γυναίκες να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους. Και θα πρέπει να αποφεύγουμε τις διακρίσεις κατά των γυναικών όταν αποκτούν παιδιά. Εγώ ανησυχώ και για την Κροατία, και για τη δημογραφική κατάσταση στην Κροατία αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Διότι ο πληθυσμός μας γυράσκει και πεθαίνει. Μια οδηγία όμως δεν μπορεί να το λύσει αυτό. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πολιτική και θα ήθελα να ακούσω κάτι τέτοιο από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε οικονομική κρίση, όμως πρέπει να θέσουμε και προτεραιότητες. Και αν στο μέλλον θα θέλαμε να έχουμε παιδιά που θα μεγαλώσουν και θα είναι φορολογούμενοι, που είναι προαπαιτούμενο για την επιβίωσή μας, θα πρέπει να το θέσουμε σαφώς σαν προτεραιότητά μας. Και αυτή η Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσουμε μέτρα προς βελτίωση της δημογραφικής καταστάσεως στην Ευρώπη που είναι καταστροφική σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ελέγχθησαν σήμερα. Προς την διακατεύθυνση ήταν όλα τα σχόλια. Δηλαδή ότι είναι απολύτως απαραίτητο να ξεμπλοκάρουμε αυτή την πρωτοβουλία οδηγίας που μετά από 6 χρόνια έχουμε μπλοκαριστεί και δεν κάναμε τίποτε. Αυτό νομίζω θα είναι το καλύτερο μήνυμα που θα στείλει η Ευρώπη για την κοινωνική της πολιτική, για να βελτιωθεί ο αέρας που αναπνέουμε όλοι. Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά τις γυναίκες, την υγεία, την ισότητα, την κοινωνική προστασία οικονομικά θέματα, δημογραφικά θέματα και νομίζω ότι αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ποιότητα ζωής ε, του μισού πληθυσμού της γης, άρα όλου του κόσμου. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το εξής. Πολλές φορές θα πρέπει να πούμε στην Προεδρία του Συμβουλίου ότι δεν είναι βραβείο το να προεδρεύει κανείς. Είναι ευθύνη είναι καθήκον και θα πρέπει να τιμήσει κανείς το θέση αυτή που του προσφέρεται και τη δυνατότητα. Η οδηγία αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και μέρος της στρατηγική μας για την οικονομική ανάκτηση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι η έλλειψη δικαιοσύνης και οι ανισότητες πάντα στην, στην αγορά δημιουργίας δημιουργούσαν ε, συνθήκες ανισότητας και οικονομικά προβλήματα και η οικονομική κρίση τι κάνει από ό,τι λέγουν. Ότι δεν επωφελούμεθα από τα προσόντα που έχει ο μισός μας ε, πληθυσμός. Ακούσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στην Ευρώπη, γι' αυτό επαναλαμβάνει ακόμη και σήμερα το Κοινοβούλιο μετά από πολλές φορές ότι είναι ευέλικτο, είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί, να συζητήσει και Έχω την εντύπωση, μιλώντας για το θέμα αυτό, ότι κάποιοι από εμά έχουν εξουθενωθεί μετά από τόσα χρόνια εργασίας και αγώνων για να φέρουμε σε πέρα στο θέμα αυτό στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Αυτό που θέλει να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που θέλει και πρέπει να ακούσει η Επιτροπή και κυρίως το Συμβούλιο είναι ότι αν η Ευρώπη έχει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει και το διαθέτει είναι για να μπορέσει τέτοιου είδου θέματα να τα κάνει να προχωρούν, διότι αφορούν δικαιώματα βασικά. Γι' αυτό παρακαλώ και για να φτάσω συγκεκριμένες παρατηρήσεις, δεν μπορεί κανείς να δουλεύει με την ε, γιλιοτίνα στο κεφάλι του ή με το ρολόι στο χέρι. Ε, υπάρχει το θέμα αυτό. Υπάρχει το θέμα του Ρεφίτ. Ας κάνουμε μια ομάδα εργασίες. Ας δώσουμε μια ευκαιρία στο Συμβούλιο να μας στείλει ένα σαφές μήνυμα, να το στείλουμε εμείς. Ας κάνουμε λοιπόν μια ομάδα εργασίας ώστε να βρούμε έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε, να μην θεωρήσουμε ότι με τέτοιε αγώνες που έχουν γίνει έχουμε φτάσει σε μια συγγενή οδηγία κάνουμε κάτι το θετικό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγητρία, στην κυρία Ρένα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω μόνο όλου του παρεμβαίνοντε και τι παρεμβαίνουσε για τι δεσμεύσει τι οποίε εξέφρασαν και την δέσμευση που είχαν αναλάβει και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Την εργασία που επιτέλεσαν στα πλαίσια τη διαμόρφωση θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και την υποστήριξη που αισθανόμαστε ότι υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε. Αυτό που ζητούμε είναι απλό. Το εξέφρασε ο συνάδελφος και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει χρόνο. Ξέρω ότι ήδη δόθηκε χρόνο, αλλά είμαστε ένα νέο κοινοβούλιο. Έχουμε και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντί μας. Έχουμε μια Προεδρία του Συμβουλίου που επίση είναι νέα. Δώστε μας χρόνο λοιπόν το χρόνο να μπορέσουμε να μαζέψουμε όλη την ενέργεια που υπάρχει για να διαπραγματευτούμε. Δεν είναι εδώ το Συμβούλιο. Νομίζω ότι προσυμφέροντο θα ήταν να ακούσει τι έχουμε να ζητήσουμε. Δηλαδή, να θέσει επιτάπητος το θέμα αυτό και να δημιουργήσει την ομάδα εργασίας των τριών προεδριών της Ιταλικής, της Λετωνικής και της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου για να προσπαθήσουμε το θέμα αυτό και στο φάκελο αυτό να προχωρήσουμε. Δεν ζητάμε στο Συμβούλιο να λάβει θέση σήμερα, αλλά να θέσει το θέμα αυτό που είναι πρωτοαρχική σημασία στη μερίσια διάταξη. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, το είπε και η πρόεδρο είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε απέναντι στο Συμβούλιο. Έχουμε υπεύθυνου βουλευτές που αναγνωρίζουν τις δεσμεύσει πρέπει να λάβουν στα πλαίσια των ευθυνών του και θέλουν να προχωρήσουν τακτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ έχετε υπόψη σα ότι η Επιτροπή μας έχει συντάξει επιστολή προς την Λετωνική Προεδρία όπου εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν προσέρχονται στις συναντήσεις μας και στις ακροάσεις μας μιλούμε για την αναγκαία συνεργασία και μάλιστα θέλουμε και working group του τρίο, το δυνατόν συντομότερο. Βέβαια το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, δηλαδή το υπαριθμό 12. Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση, αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα ήθελα δε να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μόνικα Βάνα. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι το σημαντικό αυτό θέμα ωστόσο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα άλλα. Ας περιμένουμε λίγο γιατί γίνεται πολύ θόρυβος και δεν ακούω τη φωνή μου. Ναι, ναι, θα περιμένουμε λίγο μέχρι να αποχωρήσουν οι κυρίες. Very interesting questions, Mr. Yes, yes, yes. Colleagues, we continue our uh, meeting, so please... Σας παρακαλώ, κυρία Βάνα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι που μπορώ, αγαπητές συνάδελφοι, να σας αναπτύξω την πρώτη μου γνωμοδότηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαια και νέα Ευρωβουλευτής για το θέμα πράσινη απασχόληση και αξιοποίηση του δυναμικού της πράσινης απασχόλησης για ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην αγορά απασχόλησης. Μπορώ λοιπόν να συμβάλλω και εγώ με τη γνωμοδότησή μου. Σημαντικός στόχος της γνωμοδότησης Επιτροπής μας, γιατί την έκθεση την κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης, είναι να τονιστεί το gender aspect, η πτυχή της ισότητας των φύλων δηλαδή, στις επενδύσεις για το μέλλον της απασχόλησης και να εξασφαλιστεί ώστε οι γυναίκες να ωφεληθούν με το ίδιο μέτρο στην πρόσβασή τους σε πράσινες θέσεις εργασίας, green jobs. Αυτό το περιλαμβάνω στη γνωμοδοτησή μου. Δεν υπάρχει και κανένας ενιαίος ορισμός πανευρωπαϊκής ισχύως ας πούμε για το τι σημαίνει πράσινη απασχόληση ή πράσινες θέσεις απασχόλησης Υπάρχει μια αδιαφανής μάλιστα και καμιά φορά και αντιφατική ε, κατάσταση απόψη στατιστικών δεδομένων των χωρών μελών και τα γνωρίζετε και εσείς αγαπητές συνάδελφοι ότι μια στέρεα βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για να μπορέσει να μιλήσει κανείς όχι μόνο για την συμμετοχή των γυναικών ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, δηλαδή για την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και για να μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Έτσι λοιπόν για να αναπτυχθεί ένας ενιαίος ορισμός, εγώ κάνω μια πρόταση στην γνωμοδότησή μου, να αντιχθεί υπόψη δηλαδή ο ορισμός που δίνει η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, καθώς και τα Ενωμένα Έθνη. Green jobs as decent jobs, δηλαδή αξιοπρεπείς πράσινες θέσεις εργασίας, μέσα στα πλαίσια δηλαδή τη απασχόληση που έχει σχέση με το περιβάλλον. Αυτό θεωρώ ότι από την άποψη των γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Επίση, να υπάρχει μια ενιαία θέση σχετικά με του τομεί που περιλαμβάνονται στι δραστικές. Εγώ προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση τη Βιέννη. Έχω ασχοληθεί για πολλά χρόνια με τι πράσινε θέσει απασχόληση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχαμε μάλιστα και πρόγραμμα δράσης για την πρόθεση των γυναικών σε πράσινε δουλειές στην Βιέννη είδαμε ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι για παράδειγμα και ο τομέας των δημόσιων μεταφορών ή το εμπόριο. Και αυτά δεν περιλαμβάνονται σε στατιστικά δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα εδώ χρειάζεται πρώτα-πρώτα βελτίωση των στατιστικών δεδομένων και ορισμός βέβαια της πράσινης απασχόλησης. Πριν προχωρήσω τώρα στα άλλα θέματα της γνωμοδότησής μου, έχω να προτάξω και το εξή σχόλιο. Όπως γνωρίζετε, είπα είναι η πρώτη μου γνωμοδότηση, η μεγαλύτερη πρόκληση βέβαια έγκυται στο πολύ περιορισμένο μήκος των γνωμοδοτήσεων και δεν μπορεί μέσα σε αυτά να τα περιλάβει κανείς όλα, όλες τις σκέψεις, τον προβληματισμό και τις αξιώσεις του. Κριτήριο για το τι θα περιλάβω στο γνώση του μου ήταν για μένα ότι θα περιοριστώ σε ζητήματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου. Τα ξέρετε αυτά εσείς και καλύτερα από μένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούνται τα πράγματα αυτά, αλλά έχουν, υπάρχουν και ψηφίσματα από παλαιότερα. Περιλαμβάνω μάλιστα και μερικά, ή μάλλον παραπέμπω σε αυτά, στη γνωμοδότησή μου. Και βέβαια υπάρχουν και συγκεκριμένοι προβληματισμοί που με απασχολούν από την πείρα μου και όλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα λέω αυτά για να σα εξηγήσω ποια είναι τα κριτήριά μου για την επιλογή των θεμάτων. Τώρα επί της ουσίας είπα ήδη ότι οι γυναίκες θα πρέπει να ωφεληθούν με τον ίδιο τρόπο από τις επενδύσεις σε πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και όχι μόνο, και όχι μόνο, λέω, να δημιουργούνται θέσεις υψηλών προσόντων σε τομείς όπου ούτως ή άλλως κυριορχούν οι άντρες. Αυτό το gender aspect πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη. Η έρευνα στον τομέα αυτό βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί. Το ίδιο η συστηματική συμπερίληψη των ε, φύλων σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και να εξασφαλιστεί η εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων. Επίσης, αυτά τα λέει βέβαια και η βασική έκθεση της Επιτροπής Απασχολήσεως, ο τομέας των πράσινων δεξιοτήτων Άρα ενεργητική πολιτική απασχόλησης στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι η υποστήριξη γυναικών επιχειρηματιών στον τομέα της πράσινης οικονομίας και χρηματοδότηση ιδίως μικροεπιχειρήσεων και όπως είπα βέβαια και οι κοινοφελείς υπηρεσίες καθώς και η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Αυτά όλα παίζουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να ελεγχθούν και από την ποσοτική και από την ποιοτική σκοπιά. Γνωρίζω βέβαια ότι υπάρχουν πολλοί τομεί που θα λείπουν από το κείμενό μου, από τη γνωμοδότησή μου. Ή πάντως ε, θα μπορέσω να τις στήξω μόνο περιθωριακά. Κάτι το οποίο με ενδιαφέρει όμως πολύ είναι και η προστασία της εργασίας και της ποιότητας της εργασίας καθώς και οι συνθήκες εργασίας στον τομέα της πράσινης απασχόλησης, καθώς επίσης και της εκπροσώπησης των γυναικών, καθώς και η λεγόμενη κρυστάλλινη οροφή, που δεν μπορούν να θράσουν οι γυναίκες για να ανέβουν πιο ψηλά. Και αυτά βεβαίως άπτονται και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κλπ. και ενός προγραμματισμού των πράσινων θέσεων απασχόλησης, σχεδιασμού των επενδύσεων, νέες διαθροτικές στηρίξεις και βεβαίω θα αναλυθεί υπόψη η θέση των γυναικών μέσα στην ανάπτυξη όλου αυτού του δυναμικού. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν μπορούν να περιληφθούν στη γνωμοδότησή μου λόγω των περιορισμένων σελίδων. Υπάρχει όμω η δυνατότητα υποβολή τροπολογιών. Η προθεσμία για τι οποίε, όπω είπατε και εσεί, είναι η 9η Τρίτου. Μέχρι τι 9 Τρίτου λοιπόν μπορούν να υποβάλλονται τροπολογίε που πολύ θα χαρώ να τι λάβω. Υπάρχει βέβαια και ένα meeting των Shadows και προβλέπεται η έγκριση της νομοδότησής μου για την 6η Πέμπτου, 6 Μαΐου. Ευχαριστώ κύριε Πετήρη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη γνωμοδότηση, είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, εστιάζεται στην ανάγκη συμπερίληψης των γυναικών στην δυνατότητα απασχόλησης στην πράσινη οικονομία. Η πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση πρέπει να εξασφαλίσει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακος, κάτι που σχεδιάστηκε πρέπει να συμβάλλει τους ώστε να μετακινηθεί όλη η οικονομία, όχι μόνο το τομέα των μικρομεσών επιχειρήσεων, να κινηθεί όλη η οικονομία προς το στόχο. Τα ωφέλη της πράσινης οικονομίας δεν θα πρέπει να τα απολαύσουν μόνο μερικοί αλλά όλοι και ο ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι να προφηθεί ο ρόλος των γυναικών στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας, μειώνοντας το τρόπο τις υφιστάμενες διαφορές στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο τομέα της κοινωνίας, σε ποιους τομείς οι γυναίκες σε δυσχερή θέση και μέσω παρομοίων πρωτοβουλειών πρέπει να ενισχύουμε τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Μιλώντας για γυναίκες θα ήθελα να αναφερθώ στα ενδεχόμενα ωφέλη της πρωτοβουλίας για την Ήπεθρο κυρίως για γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο. Όχι μόνο παράγουν τρόφιμα, αλλά είναι μεγάλη σημασία για τη συνοχή των οικογενειών και για τη διατήρηση της υπαίθρου και του περιβάλλοντος. Στόχος της κοινή αγροτικής πολιτικής είναι η διατήρηση της υπαίθρου και να διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της βιώσιμης ανάπτυξης υπαίθρου και οι γυναίκες, οι μητέρες είναι η ραχοκοκαλιά των οικογενειών στην Ευρώπη, κυρίως στην νοτιοανατολική Ευρώπη, οι γυναίκες παίζουν βασικό ρόλο στην προστασία της υπαίθρου και οι γυναίκες είναι σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση για διάφορους λόγους εκεί. Αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να επιφέρει βελτίωση της θέσης των γυναικών στην Ήπεθρο και καλωσορίζω τη συμπερίληψη του θέματος στην έκθεσή σας. Εκ μέρους των μελών του ΕΛΚ στην Επιτροπή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την καλή δουλειά που κάνατε και θα υποβάλουμε τροπολογίες για να καλύψουμε κάποιες συμπληρωματικές πτυχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει κυρία Ward, ευχαριστώ Μόνικα που έκανες τη δουλειά που έκανες. Είμαι υπερήφανη που σκιώδησε η εισηγήτρια. Συμφωνούμε επί πολλών πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι είναι θετικό. Αφορά το μέλλον. Το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε καλύτερη οικονομία. Καλύτερη από πλευρά συμμετοχής γυναικών, αλλά και βιωσιμότητας. Είναι μια ευκαιρία που δεν θα πρέπει να χάσουμε. Βασισμένη σε πρώτερες εργασίες της Επιτροπής Γυναικών από αυτού, έχω κάποια σημεία να τονίσω. Χρειάζεται εξοπλής εργασία, εκπαίδευση για τις γυναίκες, ε, γυναίκες επιχειρηματίες και προπτική για την ύπεθρο και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όπως λέει και η Μόνικα, η κοινωνική προπτική των πρασίνων θέσεων απασχόλησης είναι κρισίμου σημασία, διότι είναι δυσμενείς οι συνθήκες που συχνά αντιμετωπίζουν και ε, η λιτότητα έχει αντίκτυπο δυσανάλογο στις γυναίκες. Θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση, να προστατεύσουν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία, κοινωνική κοινωνικό διάλογο μεταξύ συνδικάτων και εργοδοτών. Για τι γυναίκε αυτό σημαίνει να βοηθήσουμε να ξεπεράσουν διάφορου φραγμού και να πετύχουν καλύτερη συμμετοχή των γυναικών ε, και προσλήψει των γυναικών στου πράσινου τομεί. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή κατάρτιση και παιδεία. Θέλουμε ισότιμη αμοιβή και να καλυφθούν τα κενά και διαφορέ αμοιβών θέματα υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασία που ανακαλυφθούν, αύξηση συμμετοχή των γενικών στα συνδικάτα, καλύτερη εκπροσώπηση στον τόπο εργασία του. Εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να συνε... θεωρηθεί ότι είναι συνεχώ επωφελέ για όσου εργάζονται. Πρέπει η πρωτοβουλία να ταιριάξει με την παιδεία και την κατάρτιση. Υπάρχουν διαφορετικέ εδρομέ που ακολουθούν οι ζωέ των γυναικών, να χρειάζεται επικοινόμορφη προσέγγιση στις επιστήμες, στη μηχανολογία. Πρέπει να θαρρύνουμε τις γυναίκες να μπουν εκεί από την εποχή του σχολείου. Και επαγγελματική κατάρτιση να λαμβάνει υπόψη γυναίκες, να αντιμετωπιστούν τα, οι φραγμοί που υπάρχουν, να θαρρύνουμε τις νέες να ζητήσουν να μπουν σε μαθητείες, σε προγράμματα μαθητείας, σε δυνατότητες για διαβίω εκμάθηση. Σαν γυναίκα επιχειρηματίας, επιθυμώ διακαώς να δω το επιχειρηματικό πνεύμα να σχετίζεται με τη δημιουργία πρασίνων θέσεων εργασίας και αυτό σχετίζεται με την εκπαίδευση. Πρέπει να συνοδεύονται μέχρι να μπουν σε επιχειρήσεις και να κάνουν την επιχειρήσή τους οι γυναίκες, να ανταλλάσσουν τη βέλτιση πρακτικές, η εμπειρία, καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Και το είδαμε το παράδειγμα να εφαρμόζεται στην Ασία και θα πρέπει να το κάνουμε πράσινου τομεί νέες γυναίκε επιχειρηματίες. Είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν αλλακτικά μοντέλα με συνεταιρισμού. Κοινωνικέ επιχειρήσεις, Συνεταιρισμού θέλουμε να προωθήσουν και να μην επικρατούν οι άντρε εκεί. Συνήθως η ιατρική επικράτηση ε, ταιριάζει και με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις. Αυτά και ευχαριστώ για τη δουλειά σας και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αυτό το σχέδιο κειμένου εκφράζει και πολλές ανησυχίες. Αυτές οι πράσινες θέσεις απασχόλησης, ε, διερωτώ με, ποιες είναι. Ποιες από αυτές ε, θα δημιουργούν ένα καλό περιβάλλον εργασιακό. Ποιος είναι ο πρακτικός τρόπος να περιγράψουμε την προσέγγιση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα. Οι παραδοσιακές θέσεις εργασίας που δεν πληρούν τα κριτήρια που περιγράφονται θα είναι αντικείμενο διάκρισης κατά κάποιο τρόπο. Ποιε θα είναι οι συνέπειες της πράσινη ανάπτυξη για, άλλες, ε, για άλλους τομείς της οικονομίας. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τη διατύπωση σε κάποια σημεία στη γνωμοδότηση ότι ο ρόλος της οικονομίας δεν έχει τονιστεί επαρκώς. Ίσως αυτή είναι η άποψη της εισηγήτριας και μόνο. Οι περιβαλλοντικές δεξιότητες που είναι αποφασιστική σημασίας για τη μελλοντική αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι που μου δημιουργεί ένα προβληματισμό που περιγράφω. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα όσα υπόθηκαν. Κάποιος είπε κάτι για με ποσοστίο μερίδιο, με ποσοστία συμμετοχή των γυναικών σε κάποιες θέσεις. Εμείς σαν Επιτροπή είμαστε υπεύθυνε να ρυθμίζουμε ποσοστά σε τι ποσοστό συμμετέχουν οι γυναίκες σε διάφορες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι παράλογο. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία ε, Βάνα πάλι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας, τις βρίσκω όλες πολύτιμες και χαίρομαι που θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να καταλήξουμε σε μια κοινή πορεία. Το θέμα είναι βέβαια θετικό και έχει και μέλλον. Έρχομαι τώρα στις κριτικές τοποθετήσεις σας ή και στις ερωτήσεις σας. Με συγχωρείτε να βγάλω τα ακουστικά μου. Έχω και όλα αυτά τα μαλλιά. Με ρωτήσατε για την πηγή της διατυπώσεώς μου ότι δηλαδή οι γυναίκες συχνά αγνοούνται την ε, συζήτηση αυτή. Το λαμβάνω αυτό κατά λέξη από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκα μόνη μου. Είναι διατύπωση η οποία ήδη έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και που νομίζω μάλιστα, το είπα και πριν, ότι έχει επανεληφθεί σε πολλές συζητήσεις με ειδικού, με εμπειρογνώμονες, με την κοινωνία των πολιτών και που είναι και προφανής βέβαια. Αν δείτε για παράδειγμα, η Επιτροπή των Περιφερειών τον ε, Φεβρουάριο. Αρχίζει μια πράσινη πρωτοβουλία. Λέει εκεί διάφορα πράγματα για τις γυναίκες δεν λέει τίποτα. Και πρόκειται για επίκαιρο παράδειγμα όπως αντιλαμβάνεστε που θεμελιώνει απολύτως αυτό που λέω ότι δηλαδή η οπτική της ισότητας των φύλων δεν λαμβάνεται δυο υπόψη. Τώρα, για τον ορισμό. Εγώ νομίζω ότι ένας ενιαίος ορισμός θα βελτιώσει την κατάσταση και είναι πολύ σημαντικός. Πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών επί μιας εκθέσεως της Επιτροπής Απασχολήσεως. Έτσι, αυτό είναι. Εμείς έχουμε το καθήκον να βάλουμε στην έκθεση της Επιτροπής Απασχολήσεως την πτυχή της ισότητας των γυναικών. Γι' αυτό η δική μας γνωμοδότηση θα περιλαμβάνει την πρόταση να υιοθετηθεί ένας ορισμός που να εξηγεί και τι είναι η πράσινη απασχόληση κλπ. Και βεβαίως όλα αυτά που λένε στους ορισμούς τους ο ILO, τα Ηνωμένα Έθνη κτλ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που πάμε να επινοήσουμε εμείς εδώ μόνες μας. Περιλαμβάνονται οι ορισμοί αυτοί σε άλλα ψηφίσματα άλλων διεθνών οργανισμών. Είναι όμως πια καιρός νομίζω να καταλήξουμε σε έναν ενίο ορισμό των πράσινων θέσεων απασχόλησης. Βεβαίω με μεγάλη χαρά θα συμμετάσχω και στις συναντήσεις των ε, σκιωδών εισηγητριών. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ κυρία μου, λέει η Πρόεδρος. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι μέχρι τις 9 Μαρτίου το μεσημέρι. Ένα μικρό σχόλιο να μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία για την ε, θαυμάσια συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ και πάλι. Η Πρόεδρος. Το θέμα 13 τώρα. Επένδυση για απασχόληση και ανάπτυξη. Προώθηση οικονομικής, κοινωνικής, εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Κύριε Γκρένινγκ, θα μιλήσω για λογαριασμό της Τζούλη που ε, ζητεί, ε, συγγνώμη που δεν είναι παρούσα και μιλώ τώρα σε πρώτο πρόσωπο σαν να είμαι ίδια. Ευχαριστώ την Γραμματεία για την υποστήριξή της. Ως γνωρίζετε, οι γνωμοδοτήσεις είναι σύντομες. Έτσι αναγκάζομαι να περιοριστώ στα πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για την απασχόληση. Γνωρίζω ότι αφήνω απ' έξω ορισμένα σημαντικά θέματα. Ελπίζω οι συναδελφοί μου να βάλουν επιτάπητος τροπολογίες για να συμπληρωθεί. Οι κυριότεροι τομείς που θα στοχεύσω είναι πρώτα το, η απόσταση στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις χώρες μέλη για να μην επιτρέπουν τέτοια διάκριση. Δεύτερο, η αξία που συνεισφέρουν οι γυναίκες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου δεν εκπροσωπούνται επαρκώς ως επιχειρηματίες, ως επικεφαλής μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και όμως θα ενισχυθεί η οικονομία μας αν μπορέσουν περισσότερες γυναίκες να αρχίσουν τις business. Τρίτο, γυναίκες σε, σε μερική εργασία, που είναι πιο συχνές οι απασχολήσει αυτέ για τι γυναίκες. Μάλιστα σε ορισμένες χώρε μέλη, έξι φορές παραπάνω ε, γυναίκες βρίσκονται σε μερικού χρόνου εργασία από τους άνδρες. Αυτά έχουν πολλά και σημαντικά, αυτό έχει μάλλον πολλά και σημαντικά μειονεκτήματα. Τέταρτο, η απόσταση μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων που οδηγεί σε εντονότερη αστιφιλία των ανδρών και επομένως οι γυναίκες μένουν πίσω. Αυτό μειώνει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις γυναίκες, οδηγεί όμως και σε περισσότερες οικογένειες που βρίσκονται στη φτώχεια. Τέλος, ψηφιακή οικονομία, ιδίως για το διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, που προσφέρει δυνατότητες σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο και επίσης οι γυναίκες μπορούν να εργάζονται από το σπίτι με ταχύ ίντερνετ ώστε να μπορούν να φροντίζουν καλύτερα και τα της οικογένειες. Θα συναντηθώ βέβαια με τις κύριες συγκήτριες. Αν έχετε σχόλια, πολύ ευχαρίστως να μου τα πείτε. Αυτά λέει η κυρία Τζούλι Γκέρλινγκ. Γκάμπριελ. Uh, Ευχαριστώ Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και ως σκιώδη εισηγήτρια για αυτή την γνωμοδότηση. Ως και εισηγήτρια λοιπόν για τις επενδύσεις, για τις θέσεις απασχόλησης και την αρχή, θα ήθελα να επικεντρωθώ στις θέσεις για τι γυναίκες και τις ευκαιρίε που προσφέρονται στις γυναίκες ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την ε, προσχώρησή του και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική επαγγελματική ζωή. Η συμμετοχή τους θα πρέπει να γίνει, λαμβάνοντα υπόψη ότι είναι και μέλη οικογένεια, είναι μητέρε, και δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνούμε πόσο σημαντική είναι η οικογένεια που είναι για την ε, μελλοντική δυναμικότητα της Ευρώπης πρωταρχικής σημασίας. Θέλουμε κοινωνικά να βελτιωθεί η κατάσταση των γυναικών, όπως είπε και η συγγετρία, να πληρωθούν τα κενά, να βελτιωθούν οι αμοιβές τους, και να μπορούν να μετά από την άδεια μητρότητα να επανέρχονται στι θέσει απασχόλησή του οι γυναίκε. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υποστηρικτικό για τι δραστηριότητε των γυναικών και να μπορούν να προσφέρονται θέσεις μερικής απαχώρησης και ειδική εξειδίκευσης για τις γυναίκες. Έτσι θα υποστηρίζονται και οι γυναίκες και κυρίως οι ακαδημαϊκοί γυναίκες. Ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, έχουν πρόβλημα να έχουν πρόσβαση σε θέσεις που έχουν οι συνάδελφοί τους άντρες. Η ποιότητα της, ε, των ε, δυνατήτων προσφάνειων για τη φροντίδα των παιδιών σε κάποιες χώρες είναι εξαιρετική, σε άλλες όχι. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί αυτή η ποιότητα και να είναι διαθέσιμη η κατάλληλη θέσμη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 5 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Τελευταίο θέμα, η παρούσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Γκάμπριελ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για την κατάσταση που αφορά την πολιτική κατάσταση στην, στο Αφγανιστάν, η ΑΦΕ την υπεύθυνη επιτυχία, θα ήθελα εγώ να επιμείνω στην έκθεση της ΑΦΕΣ. Πρόκειται για την πολιτική κατάσταση, την παρούσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά από τις ε, τελευταίες άμεσες εκλογές Πράγμα που σημαίνει ότι το σχέδιο γνωμοδότησης μου δεν είναι πολύ περιεκτικό. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε εγώ. Δεδομένη όμω τη έκθεση τη ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ, εγώ εστίασα την προσοχή μου στα θέματα τα οποία έχουν πιο άμεση σχέση με την παρούσα πολιτική κατάσταση και τη συμμετοχή των γυναικών όσον αφορά τη σταθεροποίηση στη χώρα αυτή. Σα καλώ λοιπόν να έχετε αυτό κατά νου όταν θα καταθέσετε τροπολογίε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε η γνωμοδότησή μας να ληφθεί πραγματικά υπόψη όταν θα γίνει η ψήφιση της έκθεσης ΑΦΕΤ. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε οξυδερκοί σε αυτά που λέμε. Ε, κατά πρώτο λόγο γίνεται λόγος εδώ για την ελεύθερη συμμετοχή των ε, γυναικών στο κοινωνικό γίγνεσθε, πρόσβαση των γυναικών στην παιδεία, στην εκπαίδευση, να μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή. Κατά τρίτο λόγο, στενή σχέση μεταξύ της πρόσβασης των γυναικών στο ε, δικαστικό ε, σύστημα και νέα ένομη τάξη και ανάγκη να ε, σταματήσει η βία κατά των γυναικών. Θα πρέπει επίση να έχουμε κατά νου ότι στην έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνονται εξή στοιχεία. Το πρόβλημα της ε, στην... όταν γεννούν οι γυναίκες. Ε, τήρηση των ε, συμβάσεων των ΟΗΕ που αφορούν οποιαδήποτε είδους διάκριση κατά των γυναικών την οποία έχει προσυπογράψει το Αφγανιστάν. Περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων, τους ευχαριστώ εκ των προτέρων, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 11 Μαρτίου αλλά ίσως υπάρξουν αλλαγές αν προβλέπετε ε, η ψήφιση της έκθεσης αυτής, ε, της νομοδότησης στην Επιτροπή μας στην συνεδρία 30 Μαρτίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μήπως μπορείτε να πείτε την άποψή σας αν το Αφγανιστάν τώρα είναι ασφαλής χώρα. Τι εννοώ. Μετανάστευση. Στην Ουγγαρία κάθε μέρα σχεδόν Έχουμε δωδεκάδες επί δωδεκάδων ανθρώπων και γυναίκες, αλλά βασικά άντρες από το Αφγανιστάν που διέρχονται τα πράσινα σύνορα όπως αποκαλούνται και υποβάλλουν αίτηση για άσυλο. Από αυτά που είπατε φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν περιστάσεις που καθιστούν τη χώρα επικίνδυνη. Υπάρχει κάτι που δεν αναφέρατε. Ποια είναι η άποψή σας. Αυτή η Επιτροπή, σαν Επιτροπή Γυναικών, πρέπει να κάνει κάποια βήματα για τη διατήρηση της ειρήνης. Προφανώς όταν μιλάμε για το Αφγανιστάν, έχουμε ειρηνευτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Μιλάμε για την ειρηνή στο Αφγανιστάν. Έχουμε κάποια ευθύνη για τις γυναίκες, εμείς σαν Επιτροπή Γυναικών. Ποια είναι η απόψή σας για την κατάσταση στην Ουκρανία, από την ίδια οπτική γωνία. Δηλαδή, ειρήνη, διαφύλαξη της ειρήνης. Ποια είναι λοιπόν η πτυχή του φίλου όσον αφορά τις προσπάθειες ε, διαφύλαξης της ειρήνης. Πρόεδρος. Δεν γνωρίζω αν θέλει συγγήτρια να αναφερθεί στο θέμα και να απαντήσει ερωτήσει, γιατί κάποιε από τι ερωτήσει σχετίζονται με την ερώτηση, όπω η Ουκρανία. Θέλετε να απαντήσετε, ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Η ερώτηση για την Ουκρανία είναι εκτό θέματο σε σχέση με τη γνωμοδότησή μου. Η γνωμοδότησή μου αφορά, όπω υπενθύμησα, την συμβολή των γυναικών για την ειρήνη στο Αφγανιστάν και ήθελα εκ νέου να επιμείνω ότι αν θέλουμε να μα παίρνουν να παίρνουμε στα σοβαρά την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που αυτή είναι πραστικά η υπεύθυνη για το θέμα, για την έκθεση. Δεν θα πρέπει να διασκορπίζουμε την προσοχή μα σε θέματα που είναι ενδιαφέροντα αλλά δεν αφορούν αυτή τη γνωμοδότηση. Σε αυτή τη γνωμοδότηση προτείνω να επικεντρωθώ επί του ρόλου των γυναικών στη σταθεροποίηση τη χώρα. Αυτό είναι ο ρόλο μα σαν Επιτροπή Γυναικών. Να πούμε ότι είναι η πρόσβαση στην παιδεία, με τα μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα και η πρόσβαση των γυναικών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων που αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ε, βιώσιμη ειρήνευση της χώρας. Αυτό αφορά την Επιτροπή μας. Τα άλλα δεν είναι ε, στην αρμοδιότητά μας. Ας μη σκορπιζόμαστε, ας επικεντρωνόμαστε επί τριών βασικών πτυχών για να μας παίρνει σοβαρά και η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Τώρα είναι ασφαλής, δεν είναι ασφαλής χώρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει μια έκθεση η οποία θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και νομίζω ότι αυτή είναι η ευκαιρία για μια ακόμη φορά θα έλεγα ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμεθα επί της υποστηρίξεως των γυναικών για την ειρήνη για να είμαστε αποτελεσματικοί. Τώρα για την Ουκρανία, η δεύτερη ερώτηση, πραγματικά δεν βλέπω τι σχέση έχει αυτή με την γνωμοδότηση είναι μια ερώτηση που όπως είπα, όπως και το θέμα για το Αφγανιστάν και τη γενική κατάσταση των γυναικών σε αυτού του είδους τη χώρα, χρειάζεται ολόκληρες εκθέσεις, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πραγματεύεται σήμερα αυτή η γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, κυρία Συγήτρια. Και τώρα θα ήθελα να ανακοινώσω την προθεσμία για τις τροπολογίες μεσημέρι τη 11 η Μαρτίου, 12 το μεσημέρι 11 Μαρτίου. Αυτά λοιπόν, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Να επενθυμίσω σε όλους ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είναι στις 5 Μαρτίου. Θα έχουμε μία-δύο εκδηλώσει για την ημέρα τη Γυναίκα 4 και 5 ε, Μαρτίου θα σας στείλουμε προσκλήσεις. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ τη γραμματεία, ευχαριστώ και του διερμηνείς. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.